δεν έχετε ιδέα τι σας περιμένει. Και την ε, ημέρα που έρχεται σας πιάνουν, δεν σας αφήνουν και ένας ενήλικας είναι έτοιμος να σας κόψει. Και σας ακροτηριάζει, πραγματικά. 200 εκατομμύρια λοιπόν κορίτσια και γυναίκες παγκοσμίω υφίστανται και είναι θύματα αυτού του εγκλήματος που κυρίως γίνεται σε μικρές ηλικίες, γύρω στα 15 είναι μια βάρβαρη πρακτική που δεν δικαιολογείται ούτε λόγω παράδοσης, ούτε λόγω θρησκείας, ούτε τίποτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει λοιπόν να καταργηθεί αυτή η πρακτική. Κάθε χρόνο όμως υπάρχουν εκατομμύρια κορίτσια που κινδυνεύουν από αυτή την απειλή. Γι' αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα πρέπει να φροντίσουμε να σταματήσει η πρακτική αυτή. Ευχαριστούμε. Χολβένι, εκ μέρους του ΕΛΚ, παρακαλώ. Πρόκειται εδώ για μια βάρβαρη πρακτική. Πολλά ήδη έχουν υποθεί και πιστεύω ότι πρωτίστως θα πρέπει να συζητήσουμε για το πόσο σημαντική είναι η πρόληψη εδώ. Με χαροποιεί το γεγονός ότι ο κύριος Σαρδένη, υπάρχει ένα πρόβλημα διερμηνίας φαίνεται. Λοιπόν, ε, ε, τα ξαναλέω από την αρχή. Αξιότιμοι συνάδελφοι, ήθελα να πω ότι πρόκειται για μια πίστευτα βάρβαρη πρακτική. Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα σχετικά απόψε και εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ σε αυτά που θα μπορούσαμε να κάνουμε στο πεδίο της πρόληψης. Η κυρία Κάνκου πιστεύω ότι ξεκίνησε μια πολύ καλή ε, πρωτοβουλία ε, και καλωσορίσαμε εδώ νεαρές κοπέλες από τη Γένεια και πραγματικά δημιουργήθηκε ένας γνήσιος διάλογος μεταξύ των γενεών. Μόνο στην Αφρική οι αριθμοί είναι σοκαριστικοί. Ε, Πάρα πολλά κορίτσια κάτω των 14 ετών έχουν γίνει θύματα αυτής της πρακτικής και πιστεύω ότι θα έπρεπε να, κάνουμε, να προσπαθήσουμε πάρα πολύ μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας με την Αφρική να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτή. Και θα πρέπει να προστατεύσουμε και να, τα κορίτσια και τις γυναίκες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε αυτές τις πρακτικές που δεν είναι καθόλου συμβατές με τη θρησκεία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε επίσης να βελτιώσουμε την κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών στον τομέα της εκπαίδευσης. Η UNESCO έχει συγκεντρώσει κάποια στοιχεία βάσει των οποίων πάρα πολλά κορίτσια στην Αφρική δεν έχουν απολύτως καμία πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτή η κατάσταση θα πρέπει να βελτιωθεί και θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία και με τις, ε, τους θρησκευτικού φορείς. Κύριος Πόλτσακ, Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ συμφωνώ με τους συναδέλφους που πήραν το λόγο πριν από μένα. Ο γενετικός ακροτηριασμός των γυναικών είναι βάρβαρη πρακτική, είναι ένα έγκλημα. Δεν ξέρω να υπάρχει καμία βάσιμη δικαιολογία παραδοσιακή, πολιτισμική. Είναι ένα έγκλημα και ντρέπομαι που στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ στη δική μας περιοχή, την πολιτιστική, είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα. Αυτό είναι πραγματικά δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Ναι, έχουμε κλειστές κοινότητες ή έχουμε νεοεισερχόμενες κοινότητες, αλλά παρόλα αυτά αυτό δείχνει ότι έχει αποτύχει η αστυνομία μας, το σύστημα δικαιοσύνης, κάτι δεν πήγε καλά. Αυτό είναι πάρα πολύ θλιβερό, πολύ θλιβερή εικόνα ε, για τον ευρωπαϊκό μας κόσμο και αξίζει καταδίκη. Πρέπει πραγματικά να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, στην πατρίδα μας και μετά να χρησιμοποιήσουμε διπλωματικούς διάβλους ούτω ώστε να πείσουμε και τους εταίρους μας σε τρίτες χώρες. Κατά την άποψή μας η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καλή, την υποστηρίζω πλήρως και όπως είπα Χρειαζόμαστε τεράστια διπλωματική προσπάθεια, ούτω ώστε να βοηθήσουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι ο γενετικός ακροτηριασμός των γυναικών και κοριτσιών είναι λάθος. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Έλενα Ντάλη έχει τώρα το λόγο. Η κυρία Πίτροπος, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Προεδρία για την συνεισφορά της στη συζήτηση. Ευχαριστώ όλους σας για τις παρεμβάσεις σας που αντικατοπτρίζουν κοινή προσπάθεια καταπολεμήσεως του γενετικού ακροτηριασμού των γυναικών. Και εγώ ενθαρρύνομαι από αυτό το γεγονός ότι όλοι μαζί είμαστε ενωμένοι σε αυτή την προσπάθεια. Θα λάβω υπόψη τις ιδέες σας, καταρτίζοντας την έστρατηγική για την ισότητα των φύλων και κατά τη διάρκεια όλων μου των εργασιών στα καθήκοντά μου ως Ευρωπαία Επίτροπο. Σας ευχαριστώ για την προσπάθεια, την αφοσίωση και την υποστήριξη του Κοινοβουλίου κατά της μάστιγας αυτής και προσβλέπω τη συνέχιση, στη συνέχιση συνεργασίας μας όπως ανέφεραν αρκετοί από εσά, αρκετά από τα αξιότιμα μέλη εδώ. Ελπίζω ότι τα εναπομένοντα έξι κράτη-μέλη θα κυρώσουν τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης προβλέπει ότι τα συμβαλόμενα κράτη πρέπει να ποινικοποιήσουν το γενετικό ακοτηριασμό ή την ενθάρρυνση ή την ε, ε, παροχή αυτής της πρακτικής. Και εγώ θα εργαστώ ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή εγω θα εργαστω ωστε η ευρωπαικη ενωση να καταφέρει να επικυρώσει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Και βασίζομαι στην υποστήριξή σας, ούτω ώστε να πείσω τα εναπομένοντα κράτη-μέλη. Και πρέπει όλοι μας να έχουμε υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια δεν θα πρέπει να περιμένουν, να μην τους αφήσουμε να περιμένουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα τελευταία ομιλήτρια είναι η κυρία του Πουράινεν αλλά πριν σας δώσω το λόγο θα μιλήσω στα αγγλικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Φιλανδική Προεδρία και ειδικά εσάς για τις προσπάθειες που καταβάλλατε για μια ε, πιο ισχυρή Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Το 2020 θα σημαδευτεί από, μια, από κάποια σημαντικά ορόσημα όσον αφορά την ισότητα των φύλων ε, όπως ε, για παράδειγμα το 25η επέτειο της ατζέντα του Πεκίνου ε, της ε, ε, ατζέντας για την βιώσιμη ανάπτυξη, την 20η επέτειο για το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών για την ε, ειρήνη και τη σταθερότητα και επίσης για την ισότητα των φύλων και το Φεβρουάριο πράγματι θα εορτάσουμε την ε, Διεθνή ημέρα μηδενικής ανοχής για ε, των πρακτικών του γυναικείου ακροτεριασμού. Κυρίες και κύριοι, ας ε, τερματίσουμε πλέον αυτή την πρακτική. Όλες οι γυναίκες και τα κορίτσια θα έπρεπε να έχουν το δικαίωμα μιας πλήρους ελευθερίας και ασφάλειας ως άτομα με πλήρη ακαιρεότητα στο Συμβούλιο της Ευρώπης τη Σύμβαση για την καταπολέμηση της γυναίκας κατά των γυναικών και οικογενειακής βίας, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δηλαδή, εκεί εκλήθηκαν όλοι προκειμένου να εξασφαλίσουν μία συνοχή μεταξύ ε, εσωτερικών και εξωτερικών ενωσιακών πολιτικών. Η καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των νεαρών κουρατσιών είναι ένα καθοριστικό στοιχείο σεβασμού των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Φιλανδική Προεδρία ε, κατέβαλε σημαντικές ε, προσπάθειες ε, στο πλαίσιο αυτής της σύμβασης και ενθαρρύναμε εκείνες χώρες μέλη που ακόμα δεν έχουν επικυρώσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης να την επικυρώσουν. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μεταξύ αυτών των ε, φορέων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει έναν ηθήνοντα ρόλο στις προσπάθειες αυτές που βρίσκονται στην καρδιά, στο επίκεντρο των κοινών ευρωπαϊκών αξιών. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και πραγματικά είναι μεγάλη μου τιμή που ολοκληρώνω τη Φιλανδική Προεδρία με αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Κύριε ε, Πρόεδρε, ε, επιτρέψατε να σας ευχαριστήσω ε, πολύ. Ήταν εξαιρετική η συνεργασία μας εδώ συζητώντας ποικίλα θέματα. Ε, πέρασα ώρες συζητώντα με τα μέλη του Συμβουλίου στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες και πραγματικά το κάθε λεπτό αυτής της συνεργασίας άξιζε τον κόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η δική μας Προεδρία φτάνει στο τέλος της, αλλά ο αγώνας για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου συνεχίζεται. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Ελπίζω όλοι να μπορέσετε να περάσετε τα Χριστούγεννα με τις οικογένειές σας και τους αγαπημένους σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση. Ε, κατά την Ολομέλεια του Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί η ψηφοφορία. Η επόμενη συνεδρίαση ε, αύριο Πέμπτη 5η ε, στις 9 έως τις 4. Ε, η μερίσια διάταξη αναφέρεται στα πρακτικά